Εξ ονόματος της Κομισιόν, ο κ. Σέτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, είναι ε, συντετριμένη για την κατάσταση στη Μαδέρα και τον υψηλό αριθμό των θυμάτων. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους κατοίκους της Μαδέρα να τους εκφράσω την ε, συμπαράστασή μου και ιδίως εις τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων. Ο Επίτροπος Ιωάννης Χάν μίλησε χθε με τον υπεύθυνο στη Μαδέρα τον κύριο Χαντίν και ε, ακούσαμε ότι η κατάσταση είναι υποέλεγχον ε, συμμετέχουν οι εθνικές και περιφερειακές δυνάμεις ε, και αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται ε, άλλος μηχανισμός ε, για την, την επίλυση της καταστροφής. Υπάρχει στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλες τις δυνατότητες για να δει ποιες χρηματικές ενισχύσεις μπορούν να δοθούν ή στην Μαδέρα, ιδίως μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή διότι σε περιφερή περίπτωση είχε δοθεί ένα μεγάλο ποσό εις ε, την Πορτογαλία. Το 2002 δημιουργήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης ακριβώς για να μπορέσει να συμπαρασταθεί στα κράτη τα οποία πλήττονται από σοβαρές φυσικές καταστροφές. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να καλύπτονται και ορισμένα κριτήρια. Εκ των, η βασικότερη προϋπόθεση είναι ε, η Πορτογαλική Εθνική Κυβέρνηση να ζητήσει βοήθεια και πρέπει να σας ε, υπενθυμίσω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, η Πομαλά Συνθήκας επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου σε μεγαλύτερες καταστροφές όταν το ποσό ξεπερνά το 0,6% του ΑΕΠ της πληττόμενης χώρας ενώ ε, εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν για την Πορτογαλία ε, καταστροφές ε, πάνω από 950 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά βέβαια σε έκτακτες συνθήκες μπορεί να δοθεί η βοήθεια αυτή και σε, για μικρότερες περιφερειακές καταστροφές για περιοχές όπως η Μαδέρα οι οποίες έχουν πληγεί. Επειδή όμως μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την έκταση της καταστροφής δεν μπορεί να αποφασίσει εάν καλύπτονται οι προϋποθέσεις αυτές. Θα πρέπει γρήγορα η Πορτογαλία να προβεί σε μία πλήρη και ε, ε, ακριβή αξιολόγηση των ζημιών και να την υποβάλει εντός 10 εβδομάδων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ο κύριος ε, Χάν έχει ήδη μεταβεί στην Πορτογαλία για να μπορέσει να συναντηθεί με τις αρχές. 6 και 7 Μαρτίου θα επισκεφθεί τη Μαδέρα για να διαμορφώσει γνώμη επιτόπου και οι αρχές ε, της ε, ε, κοινότητος θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν τις αρχές της Πορτογαλίας. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι πόροι του Ταμείου Αλληλεγγύης δεν μπορούν να διατηθούν αμέσως διότι δεν υπάρχει ένα μέσον κατεπίγουσας καλύπτεως. Χρειάζεται μία επιπρόσθετη συνδρομή των ε, κρατών μελών πέραν του τακτικού προϋπολογισμού, άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να υποβληθεί εις ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή σε εσά και στο Συμβούλιο για να κυρωθεί. Χρειάζεται δηλαδή μία μακριά διαδικασία μηνών μέχρι ότου υπάρξει αποπληρωμή. Εμείς προσπαθούμε να βραχύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις προθεσμίες αυτές. Τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν, δεν διατίθενται για τα έκτακτα μέτρα. Μπορούν να βοηθήσουν στην πιο μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξουν σύντομα συζητήσεις για αλλαγές και προσαρμογές στα προγράμματα που ενδιαφέρουν την Πορτογαλία. Πρέπει όμως να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει και τους ανθρώπους και στις αρχές στη Μαδέρα να επιλύσουν τα προβλήματα που προκάλεσε αυτή η μεγάλη φυσική καταστροφή Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα μιλήσουν οι ομάδες. Ο κύριος Τεσέιρα για... ένα λεπτό. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περνώ σήμερα το λόγο με λύπη γιατί προσωπικά είδα αυτή την τραγωδία που έπεσε πάνω στην Μαδέρα την περασμένη εβδομάδα. Και εγώ θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια αυτών των 42 θυμάτων. Η διάσταση της καταστροφής αυτής τώρα είναι ακόμα υπό Οι ερευνητικές ομάδες εργάζονται χωρίς διακοπή και μόνο τώρα φτάνουν στις πιο απομονωμένες περιοχές και μπορεί να αυξηθεί και ο αριθμός των θυμάτων. Οι ζημιές οι υλικές στις οδούς, στις υποδομές, στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι ανυπολόγιστης. 700 άτομα έχασαν την οικία τους. Η κοινωνική και οικονομική επίπτωση αυτής της κρίσης δεν αφήνει τον πληθυσμό να επανέλθει στην κανονική του ζωή. Χρειάζεται πάντως ένα μήνυμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης προς τα άτομα αυτά και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο έχουν να δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης και όταν καλείται να παρέμβουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα γιατί δεν μπορούν να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρόεδρο Μπαρόζο και τον Αμρόντιο επίτρυπο, να ε, επισκεφθούν το ταχύτερο δυνατόν επιτόπου την Μαδόηρα για να δώσουν και αυτοί ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης για την ανοικοδόμηση. Τώρα είναι ώρα να ξαναοικοδομήσουμε αυτό που η φύση μας κατέστρεψε. Αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον. Και όπως λέει και ο ύμνος της Μαδέιρα, ο πληθυσμός της Μαδέρα είναι στοικός και επιμένει. Η Μαδέρα έχει μεγάλη ιστορία και με την εργασία του θα προχωρήσει ξανά μπροστά. Ευχαριστούμε τον κύριο Τεσέρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας να διαβιβάσω τα συλληπιτήριά μας στα, θύμα, στα οικογένεια των θυμάτων και εκφράζω την αλληλεγγύη μας στον πληθυσμό που έχει πληγεί από την τραγωδία αυτή που συνέβη 20 του μηνός στην αυτόνομη περιοχή της Μαδέρα. Μεγάλη βροχή, άνεμη, κακοκαιρία άλλαξαν την όψη του Φουνσάλ και άφησαν μόνο ζημιές πίσω τους. Οι ζημίες στα δημόσια αγαθά, στις υποδομές και στις περιουσίες είναι σημαντικές. Ένα, μια πρώτη εκτίμηση, κυρία Επίτροπε, λέει ότι θα περάσουμε το 1 δις ευρώ σε ζημίες. Οπότε μπαίνουμε εντός των κριτηρίων που προβλέπει και η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Αλλά υπάρχουν και δεκάδες θάνατοι, πολύ τραυματισμένοι και αγνοούμενοι και εκατοντάδες που έχουν χάσει τις οικίες τους. Όλος ο κόσμος είδε αυτές τις εικόνες της καταστροφής. Οι εκφράσεις αλληλεγγύης προέρχονται από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσει την ενεργή της αλληλεγγύη σε αυτήν την νησιωτική και απομονωμένη περιοχή με την επίγουσα κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για να μειώσει τις ζημίες και να βοηθήσει στο να επανέρθει η ομαλότητα στην περιοχή αυτή. Και σας λέω το εξής, κύριε Επίτροπε, το Ευρωκοινοβούλιο αυτό ήδη ενέκρινε τροποποιήσεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Και αυτό γιατί, γιατί τώρα δεν ισχύουν αυτές οι αλλαγές, γιατί δεν εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ΓΟΕ, η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα ξεκινήσαμε την Ολομέλεια ε, με ενός λεπτού σιγή για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τα θύματα αυτής της καταστροφής στην Μαδέιρα και των οικογενειών τους και ένα μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους που τους βοηθούν. Όμως αυτή η ενός λεπτού συγγύη θα πρέπει να μας προβληματίσει και να προχωρήσουμε σε μια σκέψη πέραν των όσων πρέπει τώρα να κάνουμε. Στην Μαδέρα είδαμε ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς θα επαναλαμβάνεται. Οι κλιματικές αλλαγές φαίνεται ότι οδηγούν συνέχεια σε τέτοιου είδους καταστροφές. Πρέπει να αποφύγουμε τις φυσικές καταστροφές, αλλά θα πρέπει να μειώσουμε επίσης και τις επιπτώσεις του στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πολιτικές προγραμματισμού για, που, υπέρ του δημοσίου καλού. Και τελειώνω Πρόεδρε, αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν επιγόντως να αποκριθούν σε μια επίγουσα κατάσταση και χρειάζονται χρηματικά μέσα και η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Πάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Μέλο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αυτή η τραγωδία που συνέβη στην Μαδέρα κατέστρεψε πολλές ζωές, δημιούργησε πολλές ζημίες και κατέστρεψε την ομορφιά μιας πολύ όμορφης νησιωτικής περιοχής. Κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος για την βιαιότητα, την εικόνα που είδαμε και είδαμε ότι το νερό παρέσυρε σπίτια, αυτοκίνητα, γέφυρες, άλλαξε όλη η φύση από αυτή τη φυσική καταστροφή. Αυτή η τραγωδία δεν είναι μόνο που έγινε μια τραγωδία μιας περιοχής της Πορτογαλίας είναι μια τραγωδία που έπεσε πάνω σε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει και τις οικογένειες των θυμάτων και για να διορθώσουμε τις ζημίες μετά από αυτή την καταστροφή. Πρόεδρε, εδώ αναφέρθηκε ότι ο ύμνος της Μαδέιρα οδηγεί προς, την, ε, προς τα εμπρός. Όμως και ο εθνικός ύμνος της Πορτογαλίας τα ίδια λέει και πάντα πρέπει να προσπαθούμε να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες. Για άλλη μία φορά θα συμβεί αυτό και αυτή τη φορά και με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέλ για ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βεβαίως δεν είναι μια ευτυχής συγκυρία να συζητάει κανείς για αυτή την καταστροφή στη Μαδέρα και θα πρέπει να συμπαρασταθούμε στις πληγήσεις οικογένειες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει. Η αλληλεγγύη όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται εδώ και θα ήθελα εδώ να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το Ταμείο Αλληλεγγύης και θα ήθελα να δώσουμε το μήνυμα και στο Συμβούλιο να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να υπάρξει μία αναθεώρηση ε, του Ταμείου Αλληλεγγύης που το Κοινοβούλιο ζήτησε ήδη προ δύο ετών για να μπορέσει να υπάρχει μια πιο γρήγορη ε, βοήθεια εις ε, της πληγήσεις περιοχές. Η Μαδέρα τα τελευταία χρόνια είχε πάρει μεγάλους πόρους ε, του διαρθρωτικών ταμείων ε, θα ε, λάβει και περαιτέρω τις, τα επόμενα κράτη και θα πρέπει να μπορέσει να απαλύνει στο μέλλον τις επιπτώσεις αυτών των φυσικών καταστροφών. Αυτό πρέπει να επιτύχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μαδέρα και σε όλες τις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα ένα λεπτό. Πρόεδρε, η διάστηση αυτής της καταστροφής στην Μαδέρα απαιτεί να λάβουμε επίγοντα μέτρα και εξαιρετικά οικονομικά μέτρα στήριξης αυτής της αυτόνομης περιοχής με σκοπό την διόρθωση των υποδομών που έχουν καταστροφεί και θα πρέπει επίσης να διατεθούν κονδύλια για τα, τον πληθυσμό που έχει πληγεί από αυτήν την καταστροφή είναι μεγάλη η τραγωδία και συχνά όποιος έχει τα πιο λίγα χάνει και τα περισσότερα. Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε στο μέτρο του δυνατού όλους όσους έχασαν μέλη της οικογένειας τους, έχασαν τα σπίτια τους ή την εργασία τους. Τα όσα έγιναν στη Μαδέρα μας δείχνουν τη σημασία να ενισχύσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την πρόληψη των καταστροφών. Χρειάζεται λοιπόν ένα κατάλληλο οικονομικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιεί την πολιτική συνοχή ανάπτυξης υπαίθρου περιφερειακής πολιτικής για να την βοηθηθούν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του πληθυσμού, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Ευχαριστούμε. λεπτά, η κυρία Κύριε ε, Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τη Μαντεδέρα και να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας προς το λαό της. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες για το λαό, ιδίως αυτοί οι οποίοι έμειναν άστεγοι και γι' αυτό ζητούμε την Ευρωπαϊκή Συνδρομή και την αρρωγή του Ταμείου Αλληλεγγύης, πράγμα το οποίο θα βρει σύμφωνο στους πάντες. Θα πρέπει η Επιτροπή να ε, εξετάσει και να δει πώς τα ευρωπαϊκά ε, ε, προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται μπορούν να προσαρμοστούν να λάβουν υπόψη και αυτό το θέμα. Διότι υπάρχουν περιορισμοί, διότι το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έχει υιοθετήσει μία πρόταση η οποία το 2006 ε, υπερψηφίστηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλο λοιπόν τις προσπάθειες που γίνονται για μία διεύρυνση της ε, βοήθεια σε περίπτωση ε, των ε, φυσικών καταστροφών δεν μπόρεσε από το Μάιο του 2006 το Συμβούλιο να συμφωνήσει στην εφαρμογή αυτών των αρχών. Χρειαζόμαστε ένα ταμείο αλληλεγγύης το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να μπορεί να βοηθήσει τις χώρες που πλήττονται από καταστροφές. Γι' αυτό και ζητώ να υπάρξει μία αναθεώρηση του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χούμπνερ. Πάμε στο Κατσδιάι. Ο κύριος Ρούμπικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Βιλαλκουάντρας, κυρίες και κύριοι. Ε, το η ατυχία ε, είναι μία επίπτωση της ε, ε, θέρμανσης της ατμόσφαιρας και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει επίσης να επιλύσουμε. Δεν πρέπει δηλαδή μόνο να σκεφτούμε το θέμα αυτό αλλά μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε και από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους ανθρώπους της Μαδέρα που έχασαν πολλές θέσεις εργασίες και μήπως έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανοικοδόμησή τους για να μπορέσει κανείς να προωθήσει τον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Καλό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει αν μπορεί να διαθέσει πόρους από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Η κυρία Παπαδοπούλου για ένα λεπτό εκφράζω και εγώ τη βαθύτατη θλίψη μου για τη βιβλική καταστροφή που έπληξε την περιοχή της Μαδέιρα και την αμέριστη συμπαράστασή μου στην πορτογαλική κυβέρνηση. Εύχομαι ο τραγικός απολογισμός για ανθρώπινες απώλειες και αγνοούμενους να μην αυξηθεί. Ο πλανήτης μας στέλνει σήμα SOS οι κλιματικέ αλλαγέ σε συνδυασμό με του φρενήρει ρυθμού τη χρήση γη και τη βιομηχανική ανάπτυξη μαρτυρούν πόσο ευάλωτο γίνεται το περιβάλλον. Οι καταστροφικέ πλημμύρε στη Γερμανία παλιότερα, σε χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη και οι πυρκαγιέ στην Ελλάδα έχουν αφήσει ακόμη ανοιχτέ πληγέ οι καταστροφέ σίγουρα δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. ζητώ λοιπόν από την ευρωπαϊκή επιτροπή να ανταποκριθεί θετικά στι εκκλήσει του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για ενεργότερη δράση σε κοινοτικό επίπεδο για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και των επιπτώσεών του. ζητώ επίση άμεση στήριξη των θυμάτων τη μαδέιρα. είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αποτελεσματική κοινοτική πολιτική και ειδική έκτακτη χρηματοδότηση και δέσμη μέτρων για άμεση αποκατάσταση στα ζημιών χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα συλληπιτήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων. Ευχαριστώ κυρία Παπαδοπούλου. Ο κύριος, η κυρία Έτιγκερ. όλα τα θύματα στην Μαδέιρα χρειάζονται την υποστήριξή μας και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Το μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας προς τον πληθυσμό της Μαδέρα μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή απαιτεί γρήγορες διαδικασίες και διαδικασίες απλοποιημένες και εξαιρετικές για να υποστηριχθούν τα θύματα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε και όλα τα άλλα δυνατά ταμεία μέσω επίγοντων μέτρων, έτσι ώστε η βοήθεια να φτάσει επιγόντως στα θύματα και να μπορέσει η Μαδέιρα να νοικοδομήσει το ταχύτερο δυνατόν την πληγήσα περιοχή. Απαραίτητε όλα τα μέτρα να ληφθούν ταχύτατα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τραγικές πλημμύρες που έπληξαν την αυτόνομη επαρχία της Μαϊδέρα μας θυμίζουν ότι οι φυσικές καταστροφές εξαιτία των κλιματικών αλλαγών, της έλλειψης σχεδιασμού και υποδομών και της ελλειπούς ενημέρωσης και ετοιμότητας μπορούν να εξελιχθούν σε ανθρώπινη τραγωδία όπως και έγινε θυμίζω εξάλλου ότι πριν από λίγες μέρες μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρωπίνων περιουσιών έπληξαν και άλλες περιοχές της ευρώπης όπως τη βουλγαρία αλλά και την περιοχή του εύρου στην ελλάδα. και θέλω να θυμίσω ότι η οδηγία 60 του 2007 προβλέπει ότι μέχρι το 2011 τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν προβεί σε προκατακτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμυρών για τις λεκάνες απορροής και τις αντίστοιχες παράκτιες περιοχές της επικρατείας τους. είναι χρέο μας να πιέσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις για την αφομοίωση της συγκεκριμένης οδηγίας ενέργεια από τα κράτη μέλη. είναι όμω και χρέο τη ευρωπαϊκή ένωση και σε αυτό νομίζω δεν διαφωνεί κανεί να αναπτύξει ακόμα πιο έντονη και ισχυρή δράση στον τομέα πρόληψη φυσικών καταστροφών στην προστασία εν τέλει των ανθρωπίνων ζώων. Ευχαριστώ κύριε Ο κύριος Περίο. Ευχαριστώ για πυρκαγιές, άλλες για ξηρασίες, άλλες για κατολιστήσεις σαν κι αυτές. Καταραμένη πια έχει γίνει η κατάσταση στην Ευρώπη για να αποδειχθεί η κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικός ο αγώνας κατά των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει όμως τώρα πρώτα απ' όλα κατεπηγόντως να βοηθήσουμε τη Μαδέρα. και η νέα Κομισιόν να δράσει χωρίς να καθυστερήσει. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι είναι αλληλέγγυα κοντά στους πολίτες, κυρίως σε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Λοιπόν, εξ ονόματος των Ισπανών Σοσιαλιστών εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Πορτογαλία και καλώ την Κομισιόν χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς τσιγκουνιές να μεσολαβήσει γενναιόδωρα για την Μαδέρα. Ο Σιν Κέλλη έχει το λόγο. Από τότε που ήμουν μικρός μου άρεσε το κέικ της Μαδέρα. Μετά όταν μεγάλωσα ανακάλυψα ότι ήταν ένα νησί. Όταν άκουσα για την καταστροφή την περασμένη εβδομάδα αμέσως σκέφτηκα τους Πορτογάλους φίλους μου. Όλοι έχουμε πληγή και εμείς στην περιοχή μας είχαμε μια τέτοια καταστροφή γύρω στα Χριστούγεννα και εγώ θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν να βοηθήσει τη Μαϊδέρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε γενικότερα και τα κριτήρια που μπορούν να οδηγήσουν στην χρήση του Ταμείου Ελληλεγγύης. Είναι πολύ υψηλό το κατόφλι για την χρήση του ταμείου αυτού. Πολλέ από αυτέ τι καταστροφέ είναι τοπικού χαρακτήρα και καταστροφικές. πρόθεσμα. πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε τη Μαδέρα και καλωσορίζω τη δήλωση τη Κομισιόν για αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Ο κύριος Πάσκα. Η ομάδα μας ε, Ευρώπη για τη Δημοκρατία επίσης εκφράζει την αλληλεγγύη της και τη συμπάθειά της προς το λαό της Μαδέρα και ελπίζω ότι η βοήθεια θα μπορέσει να προσφερθεί πιο γρήγορα από ό,τι στην ΑΕΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πορτογαλική κυβέρνηση θα μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα στη φυσική καταστροφή της Μαδέρα. Συμφωνώ με αυτούς οι οποίοι ζητούν ένα μηχανισμό ο οποίος θα βελτιωθεί για να μπορέσουμε να αντιδρούμε στις φυσικές καταστροφές και να προσφέρουμε γρήγορα συνδρομή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλβες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και εγώ θέλω να δηλώσω εδώ την αλληλεγγύη μου για όλες τις οικογένειες των θυμάτων στην καταστροφή αυτή στην Μαδέρα. Εγώ είμαι από τις Αζόρες, είμαι Πορτογάλος και Ευρωπαίος και καλώ το Κοινοβούλιο και την Ένωση για να εκφράσουν την ενεργή τους αλληλεγγύη υπέρ της Μαδέρα και του πληθυσμού της. Απαιτείται η παρουσία της Ένωσης σε αυτήν την περιοχή. Τώρα είναι απαιτούμενη η αλληλεγγύη της Ευρώπης και είναι σημαντικό να φανεί ότι υπάρχει. Ο κύριος Όμπερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να απευθυνθώ στις οικογένειες των θυμάτων και λέμε στην Αυστρία ότι αν είναι η βοήθεια γρήγορη είναι διπλή. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πηγές από τις οποίες θα διαθέσουμε τους αναγκαίους πόρους. Θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις και προερχόμενος από μια ορεινή περιοχή περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς στη χώρα μας έχουμε κάνει ε, λάθη. Πολλές φορές ε, ε, δεν λάβαμε υπόψη την φύση και είδα μετά με συντριβή τις καταστροφές που υπήρχαν στις παιδιάδες της Αυστρίας πριν δύο-τρία χρόνια. Ε, όταν κρίνει κανείς ε, τις φυσικές διεξόδους ε, δημιουργούμε προβλήματα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες χιονοστιβάδες στην Αυστρία και δεν ήταν δυνατόν πάντα να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και εγώ είμαι έτοιμος να συνδράμω προς αυτή την κατάσταση κατεύθυνση. Η κυρία Φερέιρα, τελευταία ομιλήτρια. Και εγώ θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με την Μαδέρα και να ζητήσω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα την Κομισιό να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να βοηθήσουν την περιοχή. Να υπογραμμίσω επίσης ότι όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους καταστροφή είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες όταν αυτή συμβαίνει σε φτωχές περιοχές. Για την περίπτωση της Μαδέρα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η οικονομική βάση πλήττεται άμεσα διότι εξαρτάται από τον τουρισμό η περιοχή και όταν η φυσική ομορφιά και οι υποδομές πλήττονται είναι ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα. Είναι πιο σοβαρά λοιπόν τα προβλήματα αυτά σε φτωχές και ορεινές περιοχές και τουριστικές περιοχές όπως είναι η Μαδέιρα. Είναι απαραίτητο όλες οι προσαρμογές και οι τροπολογίες που ζητήθηκαν να γίνουν για με το Ταμείο αλληλεγγύη να μην καθυστερήσουν άλλο γιατί πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα διότι εξαιτία των κλιματικών αλλαγών τέτοιου είδους καταστροφές θα συμβούν στις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ο Επίτροπος. Αγαπητοί ε, Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσουμε την καταστροφή στην Μαδέρα. Έχετε ε, απευθύνει μία ε, εκβάθους καρδίας έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους και αυτό είναι έτοιμη να το πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις επόμενες εβδομάδες, σε στενή συνεργασία με τις αρχές, θα μπορέσουμε να επέμβουμε. Γνωρίζουμε και πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές των ταμείων. Αν υπάρχει ευελιξία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κλείνει υπέρ των συμφερόντων της Μαδέρας. Θα πρέπει όμως να υποβληθούν ορισμένες Ορισμένε χαρτιά, ορισμένε διαδικασίες και ε, γι' αυτό ο κύριο Χάν, ο συνάδελφος επίτροπος, είναι πάντοτε στη διάθεση όλων για συζήτηση και συνδρομή λέχθη ε, ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές και οι διατάξεις του Ταμείου διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει εδώ και χρόνια μία σχετική πρόταση που στήριξε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά το Συμβούλιο είχε τότε πει ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν επρόκειτο να βοηθηθούν ή να δοθούν καλύτερες δυνατότητες. Η πρόληψη πρέπει να παραμείνει ένα βασικό σημείο της πολιτικής μας και ε, η συνοχή είναι χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους και τη διοίκηση της Μαδέρας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον, η συζήτηση έκλεισε και η ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα της εμερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση από την κυρία Βάλεαν σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα για ενεργειακές υποδρομές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα